Good afternoon. I'm Καλησπέρα. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο πρώτο αντιπρόεδρο. Δέκα λεπτά σα έδωσα για να καθίσετε, να κατασταθείτε. Αρχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μα. Κυρίσω την έναρξη τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμών. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θέλω να επωφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να καλωσορίσω εδώ μία αντιπροσωπεία μελών εθνικών κοινοβουλίων της Μιαμάρ και της Σρι που ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν τη συνεδρίασή μας. Είναι βουλευτές στις χώρες τους. Δεν έχω άλλη ανακοίνωση έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει επί των πρακτικών. Εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες μας. Έχουμε τρεις γνωμοδοτήσεις να ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Και αρχίζουμε με την πρώτη, που είναι γνωμοδότηση σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020, με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της, και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Συντάκτης νομοδότησης είναι ο κύριος Τόρβαλτς. Θέλει να πει κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Καλώς. Συνεπώς, συμβιβαστική τροπολογία... Α, όχι, πρώτα να κάνω μια δοκιμή, λέει ο Πρόεδρος, πριν αρχίσουμε καλύτερα. Ε, για να ελέγξουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε λοιπόν δοκιμαστικά για να δούμε το αποτέλεσμα. Πέρα τη ψηφοφορία της δοκιμαστικής. Ωραία. Όλα καλά. Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 με προφορική τροποποίηση του ίδιου του συντάκτη γνωμοδότησης. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. 13 υπέρ, 13 κατά και μία αποχή απορρίπτεται συνεπώς. Ίγκε, η κάρτα σας για να ψηφίσετε. Εγώ προσπαθούσα να ψηφίσω, έβαλα την κάρτα μου, αλλά δεν άναψε. Οπότε δεν ε, κατάφερα να ψηφίσω, λέει ο κύριος Βαλκάρθελ. Εντάξει, είναι σαφές. Και ελπίζω να μην νομίζετε ότι ημεροληπτό. Η κυρία Γκρέσλε έψαχνε την κάρτα της, τι να κάνουμε. 32, καταπίπτει 32. 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 34. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 15-12. Τώρα, τροπολογία... Αριθμός 1. Αιτιολογικές σκέψεις. Έτσι, 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέραστη τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 27 υπέρ 2 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη γνωμοδότηση. Είναι δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Ολμπριχτ. Κύριε Ολμπριχτ, έχετε να πείτε κάτι? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Συμβαστική αριθμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, Α, έκανα λάθο λέει ο Πρόεδρο. Τροπολογία 2. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορία. Απορρίφθηκε. 15 κατά, 13 υπέρ. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 8 έχει αποσυρθεί. Η 10 έχει αποσυρθεί. 1 καταπίπτει. Τροπολογία συμβαστική 3 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 έχει αποσυρθεί. 16 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 με προφορική τροποποίηση του συγγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και η τροποποιημένη γνωμοδότηση τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 26 υπέρ 3 κατά. Συγχαρητήρια, κύριε Όλμπριχτ. Και περνάμε τώρα στην τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα, που είναι το νοσιακό πλαίσιο μετεγκατάστασης, με εισηγητή τον κύριο Ντεπρέ. Δεν είναι εδώ ο συντάκτης νομοδότησης είναι εδώ. Α, είναι και εκεί, είναι κρυμμένος, κύριε Ντεπρέ. Έχετε να πείτε κάτι ή όχι. Εντάξει, έχουν υποθεί αρκετά για αυτό το θέμα, οπότε ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία αριθμός 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προτείνω να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες από την 66 μέχρι και την 230. Είναι κανείς κατά? Καλώς. Μαζί λοιπόν όλες αυτές. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτονται. Τροπολογία 68 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε 15-13 και μία αποχή. 69 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, 72 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άλλοι δύο να ψηφίσουν. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. 10 υπέρ, 19 κατά. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107, 108 είναι ίδιες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίθηκε 15 υπέρ 14 κατά. 119 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ίδια πλειοψηφία, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα για σιγουριά. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορία. 16-12 εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άλλοι δύο, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίθηκε 15-14. 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 160 έχει αποσυρθεί. Την έχω αποσύρει. Λέει ο πρόεδρος 190 και 191 που είναι ίδιες μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 208 και 209 που είναι ίδιες, μαζί λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 216-217 που είναι ίδιες μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 222 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, πάλι θα σας προτείνω να ψηφίσουμε μαζί τις αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογίες 12, έως και 65. Έχετε αντιρρήσει, όχι. Ωραία, ψηφίζουμε μαζί λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τώρα, λογικές σκέψεις υπόλοιπε δηλαδή τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Γιατί 14, έτσι. Άλλος ένας. Ωραία, πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 17 κατά 9 υπέρ. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 και 38 που είναι οι ίδιες ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Βλέπω διαφωνίες μεταξύ των ε, κομμάτων εδώ. Πέρας της φοφορίας απορρίφθηκε 17 κατά, 12 υπέρ μια αποχή. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 έχει αποσυρθεί, Τρία τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καλά, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν για την τροπολογία 53 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρασε τη ψηφοφορίας. 44-14 το αποτέλεσμα και δύο εποχές, οπότε απορρίπτεται. Τροπολογία 3, αιτιολογικές αναφορές, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προτείνω μαζί να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες 5, 6, 7 και 8. Σύμφωνοι, υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και τώρα την τροπομένη γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεν βλέπω να θέλουν να ψηφίσουν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Σαφώς εγκρίθηκε 25 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Ντεπρέ. Αυτά με τις ψηφοφορίες. Το σημείο 7 έχει αναβληθεί. Οπότε πέρα της συνεδρίασεις και θα τα ξαναπούμε στις 5.30 για την αποκοινού συνεδρίαση που έχουμε με την ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ. Yes, we have a lot of time to reorganize. Ναι, έχουμε αρκετό χρόνο για να τα ξαναβρούμε. Εντάξει. 5.30.